της συνεδρίασης και έτσι θα δημοσιευθεί η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει μια διόρθωση όσον αφορά την 6η ε, Φεβρουαρίου 2013 στο κείμενο που εγκρίθηκε. Σύμφωνα με το άρθρο 216 εδάφιο 4 του κανονισμού, αυτό το διορθωτικό θεωρείται ότι εγκρίνεται. Αν μέχρι σε προθεσμία 24, ετών, 24 ε, ωρών από τουλάχιστον μία ομάδα ή από 40 ευρωβουλευτές ε, δεν αμφισβητείται αυτό. Το κείμενο αυτό θα το βρείτε στην, στον ιστότοπο σε séance en Και με αυτόν τον τίτλο στα πρακτικά θα δημοσιευτεί την Τετάρτη, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω πέντε νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν